χώρα σήμερα στις 12 και το επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η Ζιμπάμπου. Σας παρακαλώ πολύ να μην ξεπερνάτε το χρόνο σας γιατί έχουμε στις 12 τις προφορίες ο κύριος Κοράο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, χρόνια τώρα η ε, Ζιμπάμπου υποφέρει από την ε, στρατιωτική δικτατορία Υπάρχουν πολλές και βίαιες επιθέσεις κατά των ανθρωπινών δικαιωμάτων. Η κατάσταση στη Ζιμπάμπουε τώρα ε, απαιτεί βελτίωση των ανθρωπινών δικαιωμάτων από τον ε, Ιούνιο έχουν ξεκινήσει πολλές διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις ε, στη χώρα. Η αστυνομία έχει χρησιμοποιήσει τη βία, έχει χρησιμοποιήσει δακρυγόνα για να τις διαλύσει και πρέπει να μην λησμονούμε ότι έχουν υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με την κυβέρνηση της Ζιμπάμπου ένα σχέδιο συνεργασίας το οποίο απαιτεί ε, και τα ανθρώπινα δικαιώματα. 534 εκατομμύρια για αναπτυξιακή βοήθεια διαθέτει στη Ζιμπάμπουε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά πρέπει να αξιοποιούνται βέβαια στους προβλεπόμενους τομείς, δηλαδή η κοινωνία των πολιτών, ανθρώπινα δικαιώματα και γεωργία. Πρέπει να προχωρήσει η Μπάμπουε προς μια ε, πλουραλιστική δημοκρατία ευημερούσα και με σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κύριε Φωτίγκα, ευχαριστώ. Ο ηλικιωμένος πέρας Μουγκάμπε, 36 χρόνια στην εξουσία. Έχει φέρει πατρονία, κλεπτοκρατία, βία, διαφθορά μαζικές διαδηλώσεις. Ε, θέλει να επανεκλεγεί όμως παρόλα αυτά. Εμείς ζητούμε την άμεση απελευθέρωση των κρατουμένων, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αμερόληπτη και ανεφόρον ε, χρησιμοποίηση της ε, ανθρωπιστικής βοήθειας και τη διοργάνωση δίκαιων δημοκρατικών εκλογών άμεσα. Ο κ. Μακάλιστερ. President ladies Πρόεδρε Ταγιάννη, αγαπητοί ε, συνάδελφοι, κύριε Επίτροπη, η κατάσταση όμως όπως ακούσαμε, είναι άκρως ανησυχητική η χώρα η οποία υποφέρει κάτω από το πολιταρχικό καθεστώς ο Μουγκάμπε εδώ και 36 χρόνια άφησε το ε, μονοπάτι της Δημοκρατίας εδώ και χρόνια. Πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές προκλήσεις στη Ζιμπάμπουε είναι τεράστιες. Από κοινού με την ξηρασία δημιουργούν όλο και πιο δυσάρεστε συνθήκε, ανισότητα, φτώχεια. Είχαμε μασικές διαδηλώσεις πρόσφατα που κατεστάλησαν βία από την αστυνομία. Αυτή η άσκηση βία στη δηλώση είναι κάτι που ε, παρατηρείται όλο και πιο συχνά. Είναι απαρόδεκτο. Επίση, απαγορεύτηκε στο Χαράρι για ένα μήνο οποιαδήποτε διαδήλωση. Εμεί σήμερα ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στι αρχέ τη Ζιμπάμπη. Το κράτο δικαίου πρέπει να επικρατήσει η ελευθερία του συνέρχεστε, του συνεταιρίζεσθε, η ελευθερία έκφραση πρέπει να προστατεύονται και να είναι εγγυημένε ελευθερίε. Καταδικάζουμε τι ε, παραβιάσει ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ζητούμε το πλήρη σεβασμό των ε, πολιτικών αστικών ελευθεριών, ιδίω εν ώψη των σημαντικών εκλογών που αναμένεται να λάβουν χώρα το 2018. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Γκέρενς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε η Ζιμπάμπουε θα είχε τα πάντα για να επιτύχει από πολιτικής, οικονομικής, κοινωνικής πλευράς αν δεν είχε ένα τεράστιο εμπόδιο που ονομάζεται Μουκάμπε που ε, λειτουργεί υπό το, ε, υπό το σλόγγαν «Είμαι, θα είμαι και όταν δεν είμαι θα είναι κάποιος την οικογένειά μου». Είναι τελείω ε, διαφθαρμένο το όλο καθεστώ. Εμεί είχαμε προτείνει κάποια μέτρα. Υπάρχουν σε αυτό το ψήφισμα. Ζητούμε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να στηριχθεί η χώρα να ενισχυθούν κινήματα που στόχο έχουν την εγκαθιδρύση της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης στη Ζιμπάμπουε. Επίσης και οι χώρες ε, της Νότιας Αφρικής θα πρέπει να βοηθήσουν για να λυθεί το αφρικανικό κατά βάση αυτό ε, πρόβλημα. Και είμαστε στο πλευρό του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, πριν από τρία χρόνια το κόμμα του Μουγκάμπε κέρδισε τι εκλογέ και έχουμε μια κυβέρνηση ενότητα. Κάποια ανάπτυξη υπήρχε. Παρ' όλα αυτά, οι μισθοί παραμένουν απλήρωτοι, απολύονται δημόσιοι και η καταστολή επανέρχεται. Πρόσφατα είδαμε να καταστέλλονται οι διαδηλώσεις. Ακτιβιστές να κλείνονται στη φυλακή και να απαγορεύονται οι διαδηλώσεις. Σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να εκπέμψει ένα μήνυμα στο λαό της Ζιμπάμπουε. Ένα σχόλιο αν μου επιτρέπετε για το ψήφισμα. Ο Μουγκάμπ και περί αυτών ε, επιβάλλουν απαγορεύσεις και τα λοιπά. Όμως νομίζω ότι δεν ε, έχει πλέον ε, κάποιο αποτέλεσμα ε, το μέτρο της επιβολής επιπλέον κυρώσεων. Ευχαριστώ. Κύριος Παντσέλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μετά από διάφορες διαδηλώσεις στη Τζιμπάουε, ο πρόεδρος Μπουγκάμπε υιοθέτησε μια πολύ αυστηρή κατασταλτική γραμμή. Ο φόβος να χάσει ο φόβο να χάσει την εξουσία τον οδήγησε στον υποβάλει ήδη την υποψηφιότητά του για προεδρικές εκλογές το 2018. Όμω είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς θα κάνει ακόμα μια θητεία που θα τον οδηγούσε στην ε, ε, ηλικία των 99 ετών στο τέλος της. Ε, ε, πρόκειται για μια χώρα που έχει πληγεί από τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 100 ετών. Ζητάμε από τη Ζιμπάμπουε να τηρήσει τις διεθνεί τη ε, υποχρεώσεις, να εγγυηθεί την ανεξαρτησία του δικαστικού και να αφήσει ελεύθερε τις ε, διαδηλώσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσέξει αυτή την ευαίσθητη φάση επιμένοντας ε, στο να μην υποστούν περιοριστικά μέτρα οι άνθρωποι που είναι αντίθετοι με το καθεστώς του Μογκάμπε. Ε, θα πρέπει να γίνει μια αλλαγή στην πολιτική που θα προστατεύει τους πολίτες και θα σέβεται τις δημοκρατικές αρχές και το κράτος δικαίου. Merci, Monsieur le Président. Κύριε Φερζιά, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι η πρώτη φορά που εδώ μιλάμε για τη Ζιμπάμπουε. Ο πρόεδρος Ρομπέρ Μουγκάμπε είναι από το 80 στην εξουσία. Είναι 92 ετών. Ήδη ε, υποψήφιος για επανεκλογή. Σίγουρα πρέπει να υπογραμμίσουμε την κατάσταση στη χώρα. Η απόφαση του δικαστηρίου ε, για την, ε, σε σχέση με την ε, απόφαση του, την απαγόρευση των διαλύσεων του ΚΑΠΕ είναι ένα δείγμα. Θα πρέπει να επιτρέπονται ειρηνικέ διαδηλώσει. Αλλά πρέπει να δούμε και τι ε, οικονομικέ και τι κοινωνικέ αιτίε. Το 80% κάτω από το κατόφλι τη φτώχεια. Το 80% του ΑΕΠ στην ε, αποπληρωμή του χρέου. Σε μια χώρα που είναι ρέκορντμαν παγκόσμιο ε, και είναι και πιο διαφθαρμένη χώρα. Όταν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει αναπτυξιακή βοήθεια, θα πρέπει να μπορεί να εφαρμόζεται και η αρχή της ίχνηλασιμότητας. Ε, Επίσης, θα πρέπει οι προσπάθειες της διεθνού κοινότητας να πηγαίνουν στον πληθυσμό και ιδίω στις γυναίκες, το 68% των οποίων είναι, ε, είναι θύματα βίας. Ευχαριστώ. Επανειλημμένα μιλάμε για τη Ζιμπάμπου. Πέρυσι μας ανησυχούσε ο τρόπος με τον οποίο ε, παρανοχλούνται οι υπερασπιστές ε, του δικαίου καθώς και οι σοσιαλιστές αλλά και μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Σήμερα καταδικάζουμε ότι βία των τελευταίων μηνών είναι αλήθεια ότι έγιναν περισσότερες διαδηλώσεις. Οι πολίτες της Ζιμπάμπου έχουν ένα σωρό λόγους για να διαμαρτύρονται εξάλλου. Διαφθορά, κακοδιαχείριση, φτώχεια λόγω της ε, ε, ξηρασίας αλλά και ε, το κυνήγι των ε, ορυκτών. Σχεδόν 35 χρόνια βασιλεία στο Μουγκάμπε και κατάληξη είναι μια τελείως καταστραμμένη χώρα. Καταγγέλουμε αυτή την κατάσταση και καλούμε αλλαγή, για αλλαγή, για μια μετάβαση πολιτική που θα βασίζεται σε ελεύθερε και σωστέ εκλογέ μέσα στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτου δικαιού. Είναι η μόνη επιλογή για τη Ζιμπάμπwe. Η κυρία Κέγκε, σα ευχαριστώ. Οπότε χρειάζεται και αν χρειάζεται, θυμίζω στις αρχές της Ζιμπάμπου το περιεχόμενο της συμφωνίας του, άρθρου 97 της συμφωνίας του Κοτονού και τις υποχρεώσεις που απαραίουν από αυτό το άρθρο όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου. Ε, και μάλιστα εκφράζω τη λύπη μου για τις περιοριστικά μέτρα που έχει λάβει ο πρόεδρος Μουγκάμε που έχει αναλάβει την εξουσία από το 80. Ε, δεν μπορούμε να ανεχθούμε πλέον τη βία με την οποία διεξάγουν συστηματικά την καταστολή οποιασδήποτε ε, αντίθετη φωνής οι δυνάμεις της τάξης στην χώρα. Αυθαίρετες συλλήψει, βία κατά των γυναικών, εξαφανίσει και αυθαίρετε δολοφονίε. Ζιμπάμπουες. Ο λαός της Ζιμπάμπουε απαιτεί την δημοκρατική μετάβαση που θα βασίζεται σε ελεύθερες εκλογές, στην αλλαγή των, εξου, των, εξουσιών και είμαστε στο πλευρό σας για να στηρίξουμε τον πολιτικό διάλογο με τις αρχές και για να καταγγείλουμε κάθε παραβίαση των ε, δημοκρατικών αρχών. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ ο κύριος Μπέλντερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε τα κατασταλτικά καθεστώτα συνήθως από, ξεσκεπάζονται από μόνο τους και αυτό το, ιστορικό, αυτό το ιστορικό θεώρημα αποδεικνύεται από μόνο του και στην περίπτωση του Προέδρου Μουγκάμπε ε, ο αγώνας για ε, επιβίωση ο, πάνω από το μισό των ε, κατοίκων της Ζιμπάμπουε τρώει μία φορά την ημέρα Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Μουγκάμπε ε, περιβάλλεται από πολυτέλεια. Η ελεύθερη πτώση είναι ε, της χώρας ε, είναι γεγονός. Ο Μογκάμπε σε δύο χρόνια θα είναι πάλι υποψήφιος για τις εκλογές του 18. Αυτό είναι απαράδεκτο κύριε Πρόεδρε. Εν τω μεταξύ ο πληθυσμός ανησυχεί πάρα πολύ για το μέλλον του. η χώρα είναι τελείως κατεστραμμένη και βαζίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη. Ο κύριος Όμπερμαϊερ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Όταν ανέλαβε πριν από δεκαετίες την εξουσία στη χώρα ο Μπουγκάμπε, τον χαιρέτησαν όλοι ως μεγάλο απελευθερωτή, ε, ως φορέα δημοκρατίας ε, και Δυστυχώς ακολούθησαν ρατσιστικές επιθέσεις ε, δια της βίας αφαίρεση των γεών από τους γεωκτήμονες, διαφθορά, νεποτισμός και έτσι αυτό το πλούσιο κάποτε κράτος έγινε φτωχό, χωρίς κανένα σεβασμό ανθρωπινών δικαιωμάτων, χωρίς παραγωγή. Με υποστήριξη μόνο της διαφθοράς. Αυτό πράττουμε τώρα και εμείς το διαιωνίζουμε. Ευχαριστώ πολύ. Με το ψήφισμα αυτό καταψηφίσουμε την αιμοσταγή δικτατορία του Μουγκάμπε και αποστέλουμε ε, ένα σαφές μήνυμα στον λαό της Ζιμπάμπουε. είναι πολύ σοβαρή κατάσταση με τις παραβιάσεις των ανθρωπινών δικαιωμάτων, τις διαδηλώσεις που καταστέλλονται βία και την ε, επιρροή που έχουν οι κρατικές αρχές, κυρίως αστυνομικέ στη δικαιοσύνη. Έχουν απαγορευτεί μάλιστα διαδηλώσεις παντός τύπου ε, που ήθελαν να οργανώσουν 18 διαφορετικά κόμματα αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται κατά της διαφθοράς υπέρ της δημοκρατίας οργανώνονται μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η απάντηση κυβέρνηση ήταν να ελέγξει ακόμη περισσότερα το διαδίκτυο. Θα είναι απαραίτητο πάντως να φτάσει η επιστηστική βοήθεια σε εκείνους που την έχουν ανάγκη. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, έχουμε ήδη συζητήσει και περιγράψει την κατάσταση στη Ζιμπάμπουε. Το άρθρο 7 είναι το πιο σημαντικό για μένα σε αυτό το ψήφισμα, εκεί που γίνεται λόγος για την πρόορη κατάργηση των ε, κυρώσεων και όπου καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαναφέρει δεδομένη της ε, τραγικής κατάστασης. Το να στέλνουμε 200 εκατομμύρια ευρώ στο καθεστώς του Μουγκάμπε δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά ότι το υποστηρίζουμε. Δεν πρόκειται να φτάσουν τα χρήματα σε εκείνους που τα έχουν ανάγκη. Μόνο στη στους οικείους του Μουγκάμπε και στον περιαυτών. Πέραν του και με ιδιαίτερη έφαση λοιπόν στο άρθρο 7 υποστηρίζω το ε, κείμενο αυτό, κύριο Σκαπούτο. Ευχαριστώ. Ε, η Ζιμπάμπο πέρα από όλα τα άλλα πλήττεται από τεράστια οικονομική κρίση. Λιγότερο από 2 δολάρια την ημέρα ε, χρησιμοποιεί ο καθένα. Ιδιαίτερα στι πιο εχθριακέ περιοχέ προ τον πρόεδρο Μουγκάμπε η κατάσταση είναι χειρότερη. Σύμφωνα με την ε, Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, ο Μουγκάμπε έχει πάψει έχει την συσπιστική βοήθεια ε, προ πάνω από 2 εκατομμύρια ανθρώπου που υποφέρουν από την ξηρασία επειδή είναι εναντίον του. Η βία των διαδηλώσεων κατά για την οικονομική κατάσταση δείχνει, πώς έχουν τα πράγματα. Θα πρέπει να ελέγξουμε η χρηματοδότηση που στέλνουμε στη Ζιμπάμπο να φτάνει εκεί που πρέπει. Να απαραίτητο να δουλέψουμε για μια ειρηνική μετάβαση της εξουσίας προς τη δημοκρατία και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τηλιανίδης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Προσωπικά ε, βεβαίως και συμφωνώ και συμμερίζω με τις απόψεις και ανησυχίες σας για την κατάσταση στην Ζιμπάμπουε και πιστεύω στεναρά πως αυτή η πολύ επικοδομητική, παραγωγική συζήτηση και το ψήφισμα που τη συνοδεύει είναι πολύ θετικά βήματα και είναι σημαντικά μηνύματα προς το λαό της Συμπάμπου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει πολύ μεγάλη σημασία στην ενίσχυση του κράτους δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγίως της δημοκρατίας στην Ζιμπάμπου. Και είναι και μέσα στην... το θεματολόγιο το συνταγματικό. Θέλουμε ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε την βιώσιμη ανάπτυξη και μεγέντηση η Εθνική Ενότητα δημιουργήθηκε το 2009. Έκτοτε λάβαμε μέτρα για να βοηθήσουμε τη Ζιμπάμπουε, βλέποντα βελτιώσει στον τομέα τη κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπω ήταν η έγκριση προοδευτικού συντάγματο το 2013 που συντριπτικά έγινε δεκτό από το λαό τη ε, Ζιμπάμπουε. Επίσης, τον ίδιο χρόνο είχαμε ειρηνικέ εκλογές και τρίτον είχαμε βελτίωση ε, του ιστορικού της κυβέρνηση ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σε μια κρίσιμη συγκυρία τώρα η χώρα. Βλέπουμε μια κόπωση στα οικονομικά, βλέπουμε μεγάλες κοινωνικέ ανταραχέ αναταραχές και περισσότερο βίες ε, κοινωνικές ε, διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις. Έχουμε εκφράσει την έντονη ανησυχία μας ε, για αυτές τις δηλώσεις της 13 Αυγούστου. Η ελευθερία της διαδήλωσης κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Μπαμπού όπως και η ελευθερία έκφρασης και θα πρέπει να γίνονται σεβαστές αυτές οι ελευθερίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί από όλες τις πλευρές να εξασφαλίσουν ότι αυτά τα δικαιώματα θα μπορούν οι, οι να τα ασκούν. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφωνεί με τη δήλωση του απεσταλμένου, του εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα που ζητεί οι αρχές να εξασφαλίσουν πως ε, οι παραβιάζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα θα διώκονται Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει περισσότερες πρωτοβουλίες στα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω και της αναπτυξιακής συνεργασίας, στηρίζει το δικαστικό σώμα ε, και την ε, εκλογική επιτροπή της Ζιμπάμπουε και την εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την ε, κυβέρνηση της Ζιμπάμπου και συγκεκριμένα τη φιλοδοξία της να έχει συνεργασία με τη διεθνή κοινότητα, τους διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Βέβαια, δεν αρκεί ε, το οικονομικό πεδίο. Δεν ε, θα αρκέσει αυτό αν δεν υπάρχει μια πραγματική δέσμευση για στήριξη του κράτους δικαίου και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως λέγεται και στο Σύνταγμα της χώρας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you very much, Commissioner. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Πετρούπε. Έχω λάβει 8 προτάσεις ψηφίσματος για την